Επόμενο θέμα της ημερήσια, στην διάταξη είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Δήλωση της Επιτροπής. Όπως βλέπετε τώρα κάθονται οι Επίτροποι, αλλάζουν θέσεις και καλωσορίζω εδώ τον κύριο, τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. και μόλις είναι έτοιμος θα λάβει και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλημερίζω όλες και όλους. Στη συζήτηση αυτή πριν από τη σημαντική ψηφοφορία αυτού του πολύ σημαντικού νομοθετήματος. Πέντε χρόνια μετά την ε, το κλείσιμο των Lehman Brothers το Κοινοβούλιο, οι Υπουργοί Οικονομικών και η Κομισιόν κατάστρωσαν ένα πρόγραμμα μέτρων για να δούμε τι έπρεπε να γίνει, τι μαθήματα έπρεπε να πάρουμε από αυτήν την κρίση για να μην πληρώνουν συνέχεια την ύφη οι καταθέτες και οι φορολογούμενοι και για να σταθεροποιηθεί ο τραπεζικός τομέας. Με τον ε, κύριο Ότμαν Καράς θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα single rule book που να εφαρμόζεται σε 2.200 τράπεζες της Ένωσης ως το καλύτερο όπλο κατά του κατακαιρματισμού της ενιαίας αγοράς με παράλληλο σεβασμό της ποικιλομορφία. Με τον ενιαίο αυτό μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών όπου συνεισέφεραν πολλά και ο κύριος Γκίγκολντ και η κυρία Τίσεν πηγαίνουμε παραπέρα πέρα από το προηγούμενο αυτό μέτρο και καλύπτουμε 6.000 τράπεζες με μεγαλύτερο συντονισμό υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Εχαιρετίζω εδώ και τις προσπάθειες του Προέδρου της Μάριου Δράγκη. Το νέο αυτό σύστημα διατηρεί και σέβεται την κανόνες της ενιαίας αγοράς και μπορούν όποιοι τραπεζικοί οργανισμοί θέλουν να εισέλθουν σε αυτό το σύστημα, να ενταχθούν. Βέβαια δεν χρειάζεται καμία επα, κανένας εφησυχασμός χρειάζονται ακόμη, πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά ο ενιαίος αυτός μηχανισμός είναι ουσιώδες μέτρο αλλά ε, μόνο η πρώτη φάση προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση πρέπει να συνεχίσει η εξυγίανση των τραπεζών η Τραπεζική Ένωση που είναι το πιο σπουδαίο κοινό μας πρόγραμμα από την δημιουργία του ευρώ βασίζεται στον ενιαίο μηχανισμό επίλυσης των τραπεζικών διαφορών με βάση συγκεκριμένους και προβλέψιμους κανόνες και οι τράπεζες θα πληρώνουν για τα τραπεζικά προβλήματα και όχι πλέον οι καταθέτες ή οι φορολογούμενοι. Άρα πρέπει πρώτα πρώτα να εγκριθεί η οδηγία για την επίλυση των τραπεζικών προβλημάτων και με στόχο οι ζημίες των τραπεζών να, πληρώνονται από τους μετόχους τους κατά πρώτο λόγο και δεύτερο τους καταθέτες και μόνο και όχι πλέον από τους φορολογούμενους στο σύνολό τους. Η δυσκολία βέβαια είναι πώς θα συνδυάσουμε τη νομική ασφάλεια των ε, μετόχων με κάποια ευελιξία που απαιτείται για να μπορέσουν να απορροφηθούν ευκολότερα οι ζημίες. Επειδή το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, έγινε ένας πρώτος τριμερής διάλογος τον Ιούλιο με θετικό κλίμα και χαιρετίζω εδώ την αποφασιστικότητα των δύο συνομοθετών και ιδιαίτερα του εισηγητή σας Γκούναρ Χόκμαρκ. Η συμφωνία που επετέχθη τότε είναι ουσιαστικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος. Μετά το Single Rule Book έχουμε και ως προτεραιότητα την εγκαθίδρυση, την εφαρμογή ενός ενιαίου μηχανισμού επιλύσεων των τραπεζικών προβλημάτων, εξυγίανσης με σαφείς και απλούς κανόνες που να επιτρέπουν την εφαρμογή αποτελεσματικών αποφάσεων και μέτρων που να καλύπτουν όλους τους παράγοντες της Τραπεζικής Ένωσης. Εξάλλου το bail προβλέπει ένα ενιαίο ταμείο επίσης εξυγίανσης. Οι τράπεζες θα πληρώνουν για τις τράπεζες και που θα είναι πρικοδοτημένο επαρκώς ώστε να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ουσιαστικών τουλάχιστον λειτουργιών μιας τραπέζας σε δυσκολία. Έγινε λοιπόν στις 19 Ιουλίου η πρώτη συνεννόηση. Αύριο και μεθαύριο θα συνεννοηθώ και με τους Υπουργούς Οικονομικών στο Βίλνιους. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα γιατί η συνάδελφός σας Φερέρα προθυμοποιήθηκε να γίνει η εισηγήτρια που θα ακολουθεί τις εξελίξεις αυτές. Οι πρώτες ανταλλαγές απόψεων με τα κράτη-μέλη και με εσάς μας επέτρεψαν να κάνουμε ορισμένες αποσαφηνήσεις και να έχουμε περισσότερες βεβαιότητες για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού αυτού με βάση το άρθρο 114 και τη σχετική οδηγία. Επίσης σας προσδιορίζω ότι εμείς στην Κομισιόν εδώ δεν ζητάμε περισσότερες δικαιοδοσίε. Γι' αυτό πρότεινα η Κομισιόν να παίξει τον ελάχιστο δυνατό ρόλο στο μηχανισμό αυτό εξυγίανσης που να βασίζεται κυρίως στις εθνικές αρχές που θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Επίσης διαβεβαιώσαμε τα κράτη-μέλη ότι όλες οι χώρες και οι χώρες ΟΣΤ μάλιστα και οι χώρες home και οι χώρες host θα λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Όλες οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα παίζουν ένα ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μηχανισμού αυτού. Τώρα, η διάδραση μεταξύ του μηχανισμού και των εθνικών αρχών εκτός της Τραπεζικής Ένωσης θα καθοριστούν από την οδηγία για την εξηγένση που σας ανέφερα. Όλα αυτά λοιπόν συζητιούνται και θα συζητηθούν και στις επόμενες εβδομάδες. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου και κρατών μελών, ορισμένων τουλάχιστον. <clears throat> τις διαφορές αυτές τις συζητάμε, τις ακούω, τις παρακολουθώ, αλλά ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση αποδεκτή από όλα τα μέρη, όπως έγινε και για την εποπτεία της Ευρωζώνης και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα και οπωσδήποτε πριν το τέλος του χρόνου ή μέχρι το Μάρτιο. Εδώ υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση που θα είναι ο η κύρια πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας κατά 75% χρηματοδοτείται η οικονομία από τις τράπεζες αυτή τη στιγμή στην Αλλά με ελαχιστοποίηση των κινδύνων, με όσο το δυνατόν περισσότερη σταθερότητα δηλαδή, ώστε οι τράπεζες να μπορούν πια να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας των καταναλωτών και καταναλωτριών και των επιχειρήσεων. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Uh, I would like to make one announcement. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Επίτροπο. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση λόγω της ε, απόφασης ε, τη διάσκεψη των Πρέμιων δεν θα υπάρχει μπλε κάρτα ούτε διαδικασία κατσιάη σε αυτή τη συζήτηση. Κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Γκίγκολτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την συνάδελφο Τάισεν. Είναι ένα μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα επί χρόνια οι εθνικές αρχές δεν κατάφεραν να, να αντιμετωπίσουν την κρίση και αυτό έχει σχέση με το ότι υπήρχε μεγάλη εγκύτητα μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εθνικών αρχών και το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρξει εποπτεία για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και χρειαζόμαστε μια τραπεζική ένωση που θα μας δίνει τη δυνατότητα και μιας δυνατότητας εξυγίανσης και ενός ταμείου εξυγίανσης. Σήμερα έφτασε η στιγμή που το θέμα της εποπτείας των τραπεζών έφτασε στο σημείο να ληφθούν αποφάσεις. Σήμερα όταν μιλάμε για την ε, εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι θέμα πολιτικής δύναμης και όταν υπάρχει συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας χρειάζεται και δημοκρατικός έλεγχος, ισχυρός κοινοβουλευτικός δημοκρατικός έλεγχος. Και γι' αυτό είναι αποφασιστική σημασία και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε τόσο πολύ με το θέμα αυτό γιατί θέλουμε να έχουμε ισχυρό έλεγχο. Θέλουμε να διορίζουμε τους προέδρους αυτής της νέας αρχής και θέλουμε να έχουμε την επιλογή όχι μόνο να μας παρουσιάζει χρειάζεται ένας ή ε, μία υποψήφια ε, ε, που θα πρέπει να αποδεχθούμε. Θέλουμε να διορίζουμε και τον αντιπρόεδρο που θα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα πρέπει να ελέγχουμε εάν τα πρόσωπα αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσει δημοκρατικού ελέγχου. Και τρίτον, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου σε περίπτωση που η νέα αρχή εποπτείας δεν λειτουργεί σωστά και θέλουμε ε, να υπάρχει και ο υψηλός έλεγχος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής θα ελέγχουμε τα πρακτικά της νέας εποπτικής αρχής. Ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το επαγγελματικό απόϊτο το οποίο δεν ε, παραβιάζεται, αλλά όλα τα υπόλοιπα ε, θα ελέγχονται από το Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι σημαντικό για τους πολίτες αλλά και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, μεγαλύτερη ενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν σημαίνει λιγότερη δημοκρατία, αλλά αντίθετα θα προεπλασιάζει τη δημοκρατία και τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο θα είναι ισχυρότερα από τα δικαιώματα που είχαν ε, τα εθνικά κοινοβούλια μέχρι τώρα όσον αφορά τις τράπεζές τους. Η τωρινή βέβαια λύση είναι η ε, όχι βέλτιστη λύση διότι δεν ήταν ε, η πρώτη επιλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί τώρα. Η νομισματική πολιτική δεν μπορούσε να διαχωριστεί στο βαθμό που θα το θέλαμε. Το Συμβούλιο συνεισέφερε την πορεία αυτή, αλλά ε, οι μεγάλες ασφαλιστικές ε, εταιρείες όταν συγχωνεύονται με τράπεζες δεν μπορούν να είναι αντικείμενο αυτής της ευρωπαϊκής εποπτείας. στο ε, μέλλον ε, θα έχουμε περισσότερες αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και θα είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία που θα ισχύσει για τις αποχές. Και εδώ έχουμε κάποια σημεία που πρέπει να τροποποιηθούν. Το Κοινοβούλιο θα ήθελε και η Ευρωπαϊκή Εποπτική ε, Αρχή και το νέο όργανο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί αναλογικά να μεταχειρίζεται τις τράπεζες στο μέλλον, ούτως ώστε να μην φτάσουμε ε, ε, σε ε, ισοπαίδωση των κανόνων. Τώρα θα πρέπει, περνώντας τα επόμενα βήματα της Τραπεζικής Ένωσης, να έχουμε μια εποπτεία που θα αναλαμβάνει την ευθύνη και θα υπάρχει και λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εξυγίανση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανση θα πρέπει να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατόν και εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ορίσουμε του προέδρου το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η νέα αρχή. Με αυστηρότητα και με λεπτομέρεια θα πρέπει να ελέγχουμε του ισολογισμού των τραπεζών και θα πρέπει να φροντίσουμε ο έλεγχο να είναι ενδελεχής και κατά αυτόν τρόπο μέσω του Κοινοβουλίου να υπάρχει αυτή η εποπτεία και να υπάρχει ο διαχωρισμός των πολιτικών όπως το έχουμε αποφασίσει σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Τίσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χθε ε, είχαμε τη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης ε, και σήμερα συζητάμε την κατάσταση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και φυσικά αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να αφήσουμε την κρίση πίσω μας. Έχουμε καθυστερήσει αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο επίγονται είναι τα πράγματα. Πρέπει να καταβαλούμε διπλές προσπάθειες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί η Τραπεζική Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Τραπεζική Ένωση δεν ε, είναι απλά ο ακρογωνίος λίθος για να ενδυναμώσει την ΟΝΕ αλλά θα δώσει και εμπιστοσύνη στους πολίτες έτσι ώστε να μπορούν ε, να δουν οι άνθρωποι ότι έχει νόημα να επενδύουν ε, σε αηφόρα project που δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας. Θα έχουμε την ψηφοφορία σε λίγο και αυτό σημαίνει ότι ε, δίνουμε τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι ε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή εδώ και θα πρέπει τώρα να δούμε και τους υπόλοιπους μεγάλους ε, φακέλους ε, για να έχουμε μια τραπεζική ένωση που θα έχει αναπτυχθεί πλήρως. Ε, και εγώ είμαι αρμόδια για τα υπόλοιπα θέματα. Συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, πολλά έχουν γίνει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά προς το να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία, όμως, αν τώρα θέλουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική τραπεζική υποπτία, πρέπει να ληφθούν και κάποιες δύσκολες, σκληρές αποφάσεις. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με ένα δίκαιο τρόπο, με ασφάλεια δικαίου, χωρίς κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά. Και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με την πρόταση που έχουμε εγκρίνει. Είναι μια καλή βάση. Έτσι λοιπόν, ας προωθήσουμε το Single Rule Book με εναρμονισμένη νομοθεσία, προστατεύσουμε τους καταθέτες, ας δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη δομή των τραπεζών, γιατί δυστυχώς σήμερα τα κράτη-μέλη λειτουργούν με ένα μη συντονισμένο τρόπο. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας και πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα ανθίσει. Αυτό θα το πετύχουμε αν θα έχουμε μια κατάλληλη τραπεζική ένωση. Πιστεύω ότι οι πολίτες τότε θα μας πιστέψουν ότι το αύριο θα είναι διαφορετικό από το χτες. Θα είμαστε τότε πιο ισχυροί και θα βγούμε από αυτή την τρομερή κρίση. Σας ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε τώρα με τους ομιλητές των ομάδων. Η κυρία Βορτμαν Κόλ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. αρχίζουν, ε, υπάρχουν ε, μηνύματα ανάκαμψης ε, και δίνουν κάποια αισιοδοξία στις τράπεζες. Κάποια κράτη-μέλη υπέφεραν περισσότερο από την κρίση. Κάποια κράτη-μέλη πληρώνουν περισσότερο και οι εταιρείε και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση ή χρειάζεται να καταβάλουν υψηλά επιτόκια και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας, επομένως είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, να φροντίσει για την ανάκαμψη. Ε, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη στον ρόλο εποπτείας που έχει και θα πρέπει να διασφαλίζει και την ε, λογοδοσία και θα πρέπει και έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει ε, λογοδοσία για να είναι ένα αξιόπιστο όργανο. Ευχαριστώ την ε, Μαριάν Τάισεν και τον Σβέν Γκίγκολ, του συζητητέ μα, καθώ και την ομάδα διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν. Η Τραπεζική Ένωση δεν έχει φτάσει ακόμη, δεν είναι ακόμη γεγονό. Θα υπάρξουν και άλλα εμπόδια μέχρι ότου μπορέσει ε, ο εποπτικό μηχανισμό να λειτουργήσει στην πράξη. Και όπω ήδη είπαν οι συνάδελφοι, ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό μηχανισμός εξυγίανσης και ένα ταμείο εξυγίανσης ε, θα αποτελέσουν σημαντικούς πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης. Αν βλέπει κανείς ότι οι τράπεζες ε, δεν είναι υγιείς, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής κύριε Μπαχνιέ είναι καλή για τον νέο μηχανισμό εξυγένσης και εμείς θα πρέπει ε, να καλύψουμε τις ε, ελλείψεις που υπάρχουν σε κάποιες λεπτομέρειες στις συζητήσει που θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Εμείς θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν από τις εκλογές και έχουμε τους επόμενους μήνες για να ε, καταλήξει το Κοινοβούλιο στη θέση του. Γνωρίζουμε ότι είναι πήγοντος ε, χαρακτήρα αυτό το θέμα. αλλά παράλληλα θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε τις ε, δημοκρατικές εξουσίες που είναι απαραίτητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε ο νέος ε, εποπτικός μηχανισμός ε, να λειτουργήσει από την επόμενη χρονιά και οι τράπεζες θα προσαρμοστούν ε, στα νέα αυτά, στην αυτή κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να δούμε και ποιο θα είναι υπεύθυνο, αν θα είναι η Επιτροπή, αν θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν θα είναι ε, το Eurogroup σχετικά με την ε, ποιότητα των κεφαλαίων. Γιατί ε, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασχολείται με τον έλεγχο των κεφαλαίων, αλλά θα, υπάρξει, θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της, του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Εποπτικής Αρχή. Η ανεξαρτησία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό σε αυτή την προσπάθεια ε, της Ευρωπαϊκής, Κεντρικής, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης Τραπεζών. Με αυτά τα μέτρα θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα, δίνοντας παράλληλα και εγγυήσεις στους καταθέτες η οικονομική ανάκαμψη έρχεται σιγά σιγά και αν οι τράπεζες μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους ε, θα δώσουμε μια όθηση στην ανάκαμψη. Και αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Αγαπητοί συναδελφοί, κύριε Πίτεροπε, η ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση ήταν ε, πολύ αδύναμη και καθυστέρησε πάρα πολύ. Ωστόσο, αν ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση στο τέλο αυτή τη θητεία, εμεί ε, θα έχουμε κάνει σχετική πρόοδο για την καταπολέμηση τη κρίση στο τραπεζικό σύστημα, κυρίω ε, στην Ευρώπη. Ε, ουσιαστικά δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. όταν μπαίνει σε κερδοσκοπικά παιχνίδια, τότε θέτει σε κίνδυνο όλη την επιβίωση τη κοινωνία κοινότητα. Είναι φιλελεύθερε θέσει επιτρέπουν τοξικά ε, προϊόντα να μολύνουν τι αγορέ ε, και η επιλογή να μην ρυθμιστεί. Το σύστημα αυτό ε, οδήγησε και στη μόλυνση των τραπεζών και τελικά όλο το σύστημα τέθηκε σε κίνδυνο. Έπρεπε τα κράτη να σώσουν τις τράπεζες την ίδια στιγμή που χρηματοδοτούνται από αυτές και τελικά σχεδόν οδηγηθήκαμε στο θάνατο του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστράφηκε ε, η οικονομία και πολλές θέσεις εργασίας. Ε, το να οικοδομήσουμε μια τραπεζική ενώση φαινόταν αδύνατο πριν την κρίση, τώρα αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Όμως ε, δεν θα πρέπει να χάσουμε την όφηση των μεταρρυθμίσεων. Το Κοινοβούλιο γνωρίζει πόσο επιτακτική είναι η κατάσταση, όπως και η Κομισιόν και το έχει αποδείξει εργαζόμενο πολύ γρήγορα και σοβαρά. Εμείς οικοδομούμε ένα οικοδόμημα σε πολλούς πυλώνες. Η ενιαία αγορά πρέπει ε, επίσης να είναι ενιαία και αυτός ο πρώτος πυλώνας θα ολοκληρωθεί επίσημα σήμερα όταν θα ψηφίσουμε την νομοθεσία που θέτει την έκτα στο επίκεντρο του ενιαίου συστήματος εποπτείας και θα έχουμε και την, ε, το ρόλο της ε, τραπεζικής αρχής και τη συμμετοχή των εθνικών επιθεωρητών και επίσης θα υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος όπως είναι κάτι κανονικό στη δημοκρατία όμως δεν ε, θα χρησιμεύσει το να έχουμε κοινού κανόνε όταν μία τράπεζα μπει ε, σε κρίση να πρέπει να σωθεί με χρήματα των φορολογουμένων. Ε, μία νέα νομοθεσία που θα ολοκληρώσουμε μέχρι τα τέλη του έτου θα οδηγήσει να πληρώνουν τι απώλειε ή μετοχή με την κατάλληλη ιεραρχία. Εμεί χαιρόμαστε για την πρόταση αυτή, γιατί πριν από το καλοκαίρι δημιουργήθηκε, τέθηκε η πρόταση ε, να δημιουργηθεί ένα ταμείο εξυγείωσης που να χρηματοδοτείται από όλες ε, τις ε, τράπεζες. Ξεκινούν και οι συζητήσεις για την εναρμόνιση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως αναγνωρίζουμε εδώ τις αρχές που υπερασπίζει τη δική μας πολιτική ομάδα και τα μέσα που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του 2010 διαδικασίες διαπραγμάτευσης συνεχίζονται ακόμη και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνο να γίνει υποχώρηση ενώψη διάφορων συμφερόντων. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι αποφασιστικό στο να δημιουργήσει μία νομοθεσία για τις τράπεζες που να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, που να προστατεύεται ο φορολογούμενος από τα λάθη των μετόχων και να προστατεύονται και οι πολίτες από κίνδυνους που ποτέ δεν αποφάσισαν να αναλάβουν. Ελπίζουμε ότι και οι υπόλοιπα όργανα και το Συμβούλιο θα διέπονται από το ίδιο πνεύμα, οικονομική και κοινωνική καταστροφή που συνεχίζεται κατόπιν της κρίσης του 2008 δεν επιτρέπει να διαφύγουμε αυτή της ευθύνης. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να πω ότι επιτέλους καταλήξαμε στον τερματισμό αυτού του αγώνα δρόμου τεμποδίων που είναι ένα πρώτο βήμα προς τα εμπρός και χαιρετίζω και τη Μαριάν και τον Σβέν για όλα όσα έχουν κάνει. Είναι σημαντικό το βήμα ας πούμε. Θυμηθείτε ότι όταν το Κοινοβούλιο είχαμε, είχε ζητήσει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εποπτεία το 2010 μόλις, τότε φαινόταν υπερβολικό το αίτημα δεν βλάπτει και λίγο ικανοποίηση, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας κύριε Επίτροπε, είπατε να μην εφησυχάζουμε, αλλά πρόκειται για πολύ σημαντική αλλαγή εδώ πέρα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δεν είναι πια στενά νομισματικά τα καθήκοντά της αλλά δημιουργείται μία νέα accountability οι αποφάσεις λοιπόν που θα κληθεί να λάβει η ΕΚΤ είναι πολύ σημαντικές. Έχω όμως αντιμετωπίσει και μερικές ελλείψεις. Εμείς θέλουμε να μην τίθεται το πρόβλημα ευρωζώνη μη ευρωζώνη, αλλά όσο περισσότερες χώρες μπορούν να ενταχθούν στο νέο αυτό σύστημα για να μην αναγκαστούν μετά ορισμένες να μπαινοβγαίνουν από την Ευρωζώνη. Είναι αρνητικό λοιπόν ότι δόθηκε το δικαίωμα άρνηση κυρίας σε μερικές χώρες. Όλα αυτά πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Βέβαια δεν ζούμε σε ιδεώδη κόσμο και τέλος το ψήφισμα και αυτό πολύ σημαντικό ακούσατε χθες τον Κίφερ Χόφστατ θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εγκριθεί το κείμενο αυτό πριν τελειώσει η θητεία μας. Να μην τα αφήσουμε τα πράγματα εκκρεμή γιατί ό,τι και να πούμε για την ανάπτυξη εξαρτώνται από τη δυνατότητά μας να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας όπως πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Λάμβερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι το θέμα της δημοκρατίας, δηλαδή πώς η πολιτική εξουσία μπορεί να έχει τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα που κατά τις περασμένες ε, δεκαετίες ε, ήταν ελεύθερος ε, και απαλλαγμένος από κάθε έλεγχο στο πλαίσιο της άρσης των περιοριστικών ρυθμίσεων αλλά κυρίως διότι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να τηρήσουν ό,τι υπόλοιπο κανόνων απέμενε δεν το έκαναν και τα εθνικά συστήματα εποπτείας δεν το έκαναν οι βελγικές, γερμανικές, βρετανικές τράπεζες επέτρεπαν στις τράπεζες να επενδύουν ε, στις ε, φούσκες των ακινήτων στην Ισπανία ή αλλού ε, και δεν εμπόδισαν τις τράπεζες να αναλάβουν κινδύνους επενδύοντας στα στεγαστικά δάνεια των ΗΠΑ. Δεν εμπόδισαν την Φόρτις να αγοράσει την Μπεν Άμρο. Και γι' αυτό το σημερινό αυτό βήμα είναι πραγματικά σημαντικό και αυτή τη στιγμή φτάνει αυτό το οποίο οι πράσινοι ζητούσαν εδώ και καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να υπάρχει αυτός, ε, ε, αυτό το μέτρο της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Θα έχουμε ένα καλύτερο όπλο ελέγχου κατά αυτόν τον τρόπο από ότι μέσω του συντονισμού των εποπτικών αρχών των κρατών μελών. Αποτελεί λοιπόν ένα βήμα προόδου αυτό το σημερινό ε, βήμα, αλλά υπάρχουν δύο τεστ. Καταρχήν το τεστ αξιοπιστίας, της αρχικής αξιοπιστίας πρώτα, δηλαδή όταν θα χτενίσουμε ε, τον ισολογισμό των τραπεζών, πώς θα γίνει αυτή, αυτό το τεστ. Θα γίνει πιο λεπτομερός από τα stress test που γίνονταν ε, τα περασμένα χρόνια που ήταν πολύ επιπόλαια. Αυτό θα είναι το πρώτο τεστ ε, αξιοπιστίας και μετά ε, θα γίνει το τεστ αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δούμε αν θα μπορέσει να έχει πραγματικά τη γνώση που απαιτείται και την ε, λεπτομερή εξέταση που θα απαιτείται για να έχει πραγματικό έλεγχο επί των τραπεζών. Το δεύτερο τεστ που θα απαιτηθεί και το ανέφερε και ο Σβέν και άλλοι ομιλητέ είναι ο δημοκρατικός έλεγχος. Ένα θεσμικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ε, δείχνει ότι είναι ανεξάρτητη, για να μην πούμε ότι περιφρονεί ε, τις, ε, τα άλλα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεργαστεί και θα δούμε αν θα τηρηθούν οι διατάξεις δημοκρατικού ελέγχου στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως οφείλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σβίμπουρ. Ε, σήμερα η ε, ψήφος ε, για τον μηχανισμό αυτό αποτελείται είναι το ένα μέρος, ε, όμως ε, θέλουμε να πετύχουμε και το Ταμείο Εγγύσεων και να έχουμε και ένα κοιτανό Ταμείο Εξυγίασης για τις τράπεζες που βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση. Όμως δεν πρέπει να βιαστούμε, πρέπει να έχουμε μια καλή αρχιτεκτονική για την Ευρωζώνη και ε, όλες αυτές οι προσπάθειες αφορούν όλους όσους είναι και εκτός του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τις μελλοντικές συνέπειες για όλους τους παίκτες οι ε, ασφαλιστικές δικλίδες ε, που χρησιμοποιούμε και σε εθνικό πλαίσιο έχουν διασφαλιστεί σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ανεξάρτητος επόπτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ανεξαρτησία δεν σημαίνει μη λογοδοσία. Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου έχει επιμείνει σε μια διοργανική συμφωνία που δίνει μεγαλύτερο έλεγχο του Κοινοβουλίου για τις αποφάσεις της ΕΚΤ για την εποπτεία. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα που θα σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε μια θέση να κατανοήσει και να εξηγήσει στους πολίτες τις δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να λάβει έκτη στο μέλλον για την κατάσταση των τραπεζών και την οικονομία συνολικά. Η ομάδα μου ήθελε να διασφαλίσει ότι ε, θα παραμένουν ξεχωριστά η πολιτική εποπτεία και πολιτική διοίκηση. Η πολιτική διοίκηση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την πολιτική. Χαίρομαι που έχει επιτευχθεί αυτό, γιατί ε, θα πρέπει και οι συγκεκριμένε αποφάσει εποπτεία ε, να προτείνονται για έγκριση στο Συμβούλιο. Βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο συμμετέχουν περισσότεροι από χώρε εκτό Ευρωζώνη εμεί. Ε, η δική μου χώρα δεν πρόκειται βέβαια να μπει στην Ευρωζώνη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τα μέλη τη διαπραγματική τη ομάδα και κυρίω του δύο συγητέ ε, που αναγνώρισαν ότι για να λειτουργήσει η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκε και των χωρών εκτό Ευρωζώνη. Αυτό το πακέτο που θα ψηφίσουμε σήμερα θέτει τον νέο αποπτικό μηχανισμό για την Ευρωζώνη ενώ σέβεται την ακαιρεότητα τη ε, νέα αγορά. και καθώ πολλέ τράπεζε λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιτυχία του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού είναι πολύ σημαντική για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν δύσκολο ε, για κάποιους βουλευτές να υποστηρίξουν ένα διτό τρόπο ψηφοφορίας ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Όμως ε, για τις χώρες που είναι εκτός Ευρωζώνης και αυτό αποτελεί κλειδί για τη μελλοντική οικονομική ανάκαμψη. Μεγάλα project που αποφεύγουν να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα είναι μια αιτία για την κρίση του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης και άλλοι συνάδελφοι ε, είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στα θέματα αυτά. Να δυσφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για άλλα τα κράτη-μέλη και να επιλέξουμε να μείνουν όσοι επιθυμούν εκτός του συστήματος κάνει διαφορά, αλλά κυρίως και για τους δικούς μου ψηφοφόρους. Ένα πιο ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σύστημα για την Ευρωζώνη γίνεται πραγματικότητα με μια ευρύτερη ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αναγκαιότητα μιας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και ενός Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού είναι αναμφισβήτητη και για μένα όπως και για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ε, δομείται αυτή η Τραπεζική Ένωση μου δημιουργεί αμφιβολίες. Ήδη αναφέρθηκε ότι παραμένει το πρόβλημα, ότι παραμένει περιορισμένη η τραπεζική στην Ευρωζώνη και όχι στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Παραμένει λοιπόν ε, το ζήτημα του πώς ε, θα καλυφθούν τα κενά. Παραμένει και το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συζητήθηκε πολύ στην Οικονομική Επιτροπή και στη Διαπραγματευτική Ομάδα το αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ε, ε, θα εμπλεκεί στη διαδικασία. Πιστεύω ότι είναι ε, ένα πρόβλημα που δύσκολα θα επιληθεί όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει έλεγχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επί της ε, ε, αρχής εποπτείας και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στη Διοργανική Συμφωνία και παραμένει ακόμη το ερωτηματικό για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να επιληθούν τα προβλήματα. Ε, και υπάρχουν σφάλματα το μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί. Είναι η δεύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται τώρα για ένα μηχανισμό. Πρώτος, η πρώτη προσπάθεια απέτυχε και φοβούμαι ότι και αυτή η δεύτερη προσπάθεια είναι ε, μόνο εν μέρη μια λύση. Θα οδηγήσει, ε, ε, ελπίζουμε, σε σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και ελπίζουμε ότι θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει. βασιστήκαμε στην συνθήκη της Λισαβόνας και ο κύριος Γκίγκολτ αυτό έκανε στην διαμόρφωση της έκθεσης. Παίζει όμως ρόλο εδώ και το Συμβούλιο γιατί θα πρέπει το Συμβούλιο να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε να υπάρχει μια τραπεζική ένωση όπως ζητήθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές και για να μπορέσει να εφαρμοστεί μέσα στα επόμενα χρόνια μια τέτοια τραπεζική ένωση. Ελπίζω το Συμβούλιο να γνωρίζει αυτή την ευθύνη την οποία έχει βάσει των συνθήκων και ελπίζω να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Μοργάντη. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι κατά του να έχουμε μεγαλύτερη υποπτία του τροπεζικού τομέα. Αν είχαν γίνει και κατάλληλοι αλήθεια στο παρελθόν, πιθανότατα η κατάσταση δεν θα ήταν τροστακή για πολλές τράπεζες. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο Τράκη που λείπει σήμερα, που ήταν όταν συνέβαιναν όλα αυτά ε, τα προβλήματα με την ε, μόνη την Ντιπάση και τη Σιένα, γιατί ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων ε, οφείλεται στα προβλήματα που είχε η τράπεζα των Βενετά. Όταν αγοράστηκε ο πρόεδρος Τράκη γνώριζε την αξία της Αντων Βένετα, γιατί μόνο δύο χρόνια πριν είχε εργαστεί ως ε, σύμβουλο στην Goldman Sachs. Ε, όμως ε, τότε δεν έκανε τίποτα και έγιναν κάποιες λανθασμένες αξιολογήσεις στο θέμα της τραπεζικής εποπτείας. Όμως πάντοτε το ουσιαστικό ερώτημα είναι ένα άλλο που είναι γραμμένο ότι πρέπει εξαναγκαστικά να σωθούν όλες τις τράπεζες που βρίσκονται σε δυσκολία. Θα πρέπει να παρεμβαίνουμε μόνο στην περίπτωση που έχουμε τράπεζες που που καταθέτουν οι πολίτες τα χρήματά τους, όχι σε τράπεζες που προβαίνουν σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Όλα αυτά θα ήταν δυνατά αν ε, επιστρέφαμε στο μοντέλο classical, γιατί διαφορετικά ε, έχουμε αυτό το πρόβλημα που διέπει όλες τις τράπεζες και θα έπρεπε να επιληθεί το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Ζάιλστρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι πια ανεξάρτητη και όμως ήταν ένας από τους στόχους της συνθήκης αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επομένως παραβιάζει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη. Χρηματοδοτεί κράτη. Και αυτό σημαίνει ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλες παραβιάσεις του άρθρου 132 ιδιαίτερα για την ανεξαρτησία. Η τραπεζική εποπτεία είναι κάτι που το συζητούμε πολύ αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το 11 επίσης στις Βρυξέλλες υπήρχε έλεγχος των τραπεζών, η δέξια ας πούμε. Και υπάρχουν και άλλες τράπεζες που σήμερα διαλύονται, πτωχεύουν. Πώς μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι θα τα λύσουμε όλα αυτά πανενωσιακώς. Υπάρχει εδώ ένα θέμα όχι οικονομικό αλλά πολιτικό. Και τελικά είναι χάρτινη τίγρης αυτή η εποπτεία και η ΕΚΤ. Μιλάμε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έμεσα όμως μέσω της χρήσης των χρημάτων των καταθετών Αυτά ζήτησε λοιπόν κύριε Πρόεδρε η Κομισιόν και πολλές από τις ομάδες εδώ μέσα. Δεν γίνεται, γίνονται πια σεβαστές οι συνθήκες ούτε σεβόμαστε τους πολίτες. Και του χρόνου οι πολίτες θα το δείξουν αυτό με την ψήφο τους. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τελευταίος θα ξαναμιλήσει ο Επίτροπος Μπαρνιέ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που λάβατε το λόγο. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό και όπως είπε και η συγγήτρια Μαριάν Τίσεν είναι, πρόκειται εδώ για ένα από τα κύρια θεμέλια που τίθενται με την ψηφοφορία για τη δημιουργία αυτής της Τραπεζικής Ένωσης. Οι αποταμιευτές, οι πολίτες υπέφεραν και ζημιώθηκαν από αυτή την κρίση αλλά όπως είδαμε και στο Z20 στην Αγία Πετρούπολη τελευταία ζητήθηκε παγκοσμίως μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πιο υπεύθυνος ρόλος από την Ένωση. Αυτό ακριβώς θα οικοδομήσουμε σιγά σιγά και υπομονητικά με αυτή την Τραπεζική Ένωση. Συμμερίζουμε την άποψή σας ότι πρέπει από τώρα με αποφασιστικότητα να αρχίσουμε να δημιουργούμε και το δεύτερο θεμέλιο της Τραπεζικής Ένωσης και συγχαίρω την κυρία Φερέρα και την ενθαρρύνω σε αυτά που είπε γιατί συμφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και η κυρία Γκουλάρ και ο κύριος Φερχόφστατ χθε το είπαν οι Υπουργοί Οικονομικών που θα συναντήσω αύριο στο Βίλνιους το ίδιο νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουν. Κύριε Μοργκάντη, δεν τελείωσε ακόμα ο γύρος όλων αυτών των εγγράφων και νομοσχεδίων. Υπάρχει και το θέμα του shadow banking και ένας νέος κανονισμός για τη δημιουργία benchmarks Επίσης κύριε Μοργκάντη, ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των παραδοσιακών λειτουργιών των τραπεζών και των επενδυτικών τους λειτουργιών είναι κάτι το οποίο θα το προτείνουμε ρητά ήδη από τον Νοέμβριο. Επίσης προς τον κύριο Σάριστρα θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη προσοχή και με πολλή δουλειά προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από, τις αρχικές, από τα αρχικά της καθήκοντα της ανεξάρτητης ε, νομισματικής σταθεροποίησης που είναι ο κύριος ρόλος της και του νέου της ρόλου που προβλέπει όμως η συνθήκη δηλαδή της εποπτείας. Επίσης προς την κυρία Σουίνμπον θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την απόψή της όπως και της κυρίας Γκουλάρ για τον ρόλο που πρέπει να παίζει μέσα στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού εποπτείας να παίζουν οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη αλλά που θα ήθελαν εθελοντικά να συμμετάσχουν σεβόμενες όμως την ε, ενιαία αγορά των 28 χωρών μελών. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Κύριε Λάμπερτς, μιλήσατε για την αξιολόγηση για τους λογαριασμούς των τραπεζών. Αυτό η ΕΚΤ θέλησε να το αναλάβει πριν ακόμη μιλήσει για εποπτεία. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν πολύ αυστηρά και πολύ προσεκτικά και δεν θα ήταν αδύνατον να τα κάνει αυτά ένας τρίτος ανεξάρτητος οργανισμός αλλά επίσης η ΕΚΤ πρέπει να γνωρίζει τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων και ισολογισμών για να μπορεί να παίξει καλύτερα τον κεντρικό της ρόλο. Κύριε Κλούτε, νομίζω ότι στην κλίμακα ακριβώς και των 28 χωρών πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος των ισολογισμών και με μεγάλη σοβαρότητα και αυστηρότητα. Τέλος, ευχαριστώ εκ νέου τον Σβέν Γκίγκολντ για την εργασία του ως εισηγητή και ο Φιλίπ Λαμπέρτ ανέφερε ότι οι ελεκτικές εξουσίες που είχατε ζητήσει ως κοινοβουλευτική είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο και χαίρομαι ιδιαίτερα για την τελική διαθεσμική συμφωνία μεταξύ ΕΚΤ και του Κοινοβουλίου σας, κάτι που υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο και υποστηρίζω και εγώ την θέλησή σας να παίξετε πλήρως τον δημοκρατικό σας ρόλο και ευθύνη. Βέβαια, υπάρχουν και κανόνες εμπιστευτικότητας εδώ που πρέπει να ισχύσουν, αλλά νομίζω ότι και από αυτού μπορούμε να συμφωνήσουμε για να καταλήξουμε τελικά σε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Όπως είπα και πριν δεν τελειώνει εδώ η προσπάθειά μας, δεν εφησυχάζουμε και όταν θα τελειώσει η προσπάθεια και δημιουργηθεί ο πρώτος πυλώνας ήδη από του χρόνου της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να αρχίσουμε αμέσως να δουλεύουμε για τον δεύτερο κυρία Φερέρα μου με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια θέληση να πετύχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Έληξε η συζήτηση. Και τώρα διάλειμμα μέχρι την ψηφοφορία στις 12.